της, ε, όπως επίσης και στην επερχόμενη Προεδρία. Για την περίπτωση του Δούναβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και φτάσαμε εσείως στην τελευταία έκθεση της σημερινής βραδινής συνεδρίας, που είναι η έκθεση της κυρίας Κράτσας Τσαγκαροπούλου σχετικά με τη συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης με ειδική αναφορά στο στόχο 2. Τον λόγο έχει η συγγήτρια για τέσσερα λεπτά. Το πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Ο σκοπός της έκθεσης είναι να αναδείξει τη σημασία που έχει η περιφερειακή πολιτική για την ανάκαμψη σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στον απόϊχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των επιπτώσεών της στην πραγματική οικονομία θέλουμε να τονίσουμε ότι η περιφερειακή πολιτική αποτελεί την, τη βασική πηγή επενδύσεων για την ανάπτυξη και τα διαρθρωτικά ταμεία δεν είναι μόνο εργαλεία κατάσβεσης ε, ανομαλιών και διαρθρωτικών προβλημάτων αλλά αποτελούν εργαλεία τα οποία πρέπει να προσαρμοστούν στις παρούσες συνθήκες και να αξιοποιηθούν τον καλύτερο τρόπο για την ισόρροπη ανάπτυξη για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. η έκθεση εστιάζεται ιδιαίτερα στις περιοχές του στόχου 2, περιοχές οι οποίες έχουν ε, από το 2000 ε, ήδη ε, αυξημένα ποσοστά αεπ και επίσης ιδιαίτερες επιδόσεις στην ανταγωνιστικότητα στην καινοτομία και στην έρευνα. με τη μεταρρύθμιση του 2006 οι περιοχές του στόχου 2 ε, εστιάστηκαν στην ανταγωνιστικότητα και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Σήμερα θα ε, σας έλεγα χαρακτηριστικά για να καταλάβουμε το εύρος αυτής της πρωτοβουλίας είναι 168 οι περιοχές σε 19 κράτη-μέλη της Ένωσης και αφορούν 314 εκατομμύρια κατοίκους οι παρεμβάσεις του στόχου 2 οι προσπάθειε μα λοιπόν αυτές πρέπει να συνεχιστούν σήμερα σε ευρωπαϊκό εθνικό και τοπικό επίπεδο. γίνεται σαφέ από το προτινόμενο ψήφισμα ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε την περιφερειακή διάσταση της στρατηγική για την ευρώπη του 2020 ε, μια προτεραιότητα η οποία δεν αποβλέπει μόνο στην περιφερειακή και την κοινωνική συνοχή αλλά και στην ανταγωνιστικότητα των περιοχών το ψήφισμά μας καλεί την ε, ευρωπαϊκή επιτροπή για μεγαλύτερη ευελιξία στην χορήγηση πιστώσεων και στην λήψη αποφάσεων για την καλύτερη αξιοποίηση και γρηγορότερη των διαρθρωτικών ταμείων. ήδη ε, σημειώνουμε ότι σε σύνολο 117 επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 13 τροποποιήθηκαν σε ορισμένες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσαρμόστηκαν στις συνθήκες με τις δυσκολίες τις δημοσιονομικές και τις δυσκολίες της συμμετοχής του εθνικού προϋπολογισμού. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες των χωρών μελών για να μπορέσουν να κάνουν χρήση αυτής της προσαρμοστικότητας. Η ε, βασική μας πρόταση είναι υποστηρίζουμε την απόφαση του Συμβουλίου για να ε, ενισχύσει τις προκαταβολές σε χώρες που έχουν πτώση του ΑΕΠ πάνω από 10% ή έχουν υποστήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την δημοσιονομική τους προσαρμογή και επίσης ζητούμε να ε, δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα ευέλικτων λύσεων όσο αφορά τους κανόνες νη συν 2 και νη συν ούτως ώστε τα κράτη μέλη που έχουν δυσκολίες δημοσιονομικές να μην χάσουν τις ενισχύσεις τις ευρωπαϊκές. Κάτι άλλο που επισημαίνουμε είναι ότι η έκτη έκθεση για τη συνοχή δεν δίνει αρκετά στοιχεία ποιοτικά και ποσοτικά για τις ε, περιοχές ε, του στόχου 2. Λοιπόν, ζητούμε μια μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μας δώσει όλες αυτές τις ε, απαραίτητες πληροφορίες ούτως ώστε να μπορέσουμε να παρεύουμε στην προσαρμοστικότητα στην παρούσα κατάσταση αλλά να προετοιμάσουμε και τις επόμενες δημοσιονομικές προεπτικές βάσει των πραγματικών συνθήκων και των πραγματικών αναγκών. Ε, άλλο θέμα το οποίο επισημαίνουμε είναι ότι σε ειδικέ πτώσεις όπω είναι αυτή που μας έδωσε αφορμή και για την έκθεση η οικονομική κρίση είναι αναγκαίο να καταστεί ακόμη πιο ευέλικτο ο κανόνας συν 2 λαμβάνοντα υπόψη του στόχου ε, ε, τους πολιτική στόχους της πολιτικής και τι επιπτώσει των κυκλικών οικονομικών μεταβολών στα δημόσια οικονομικά και στι ιδιωτικέ επενδύσει. Επίση, επισημαίνουμε την σημασία που έχει η προώθηση των πρωτοβολιών Jaspers, Jeremy, Jessica, διότι υπάρχουν χώρες όπως η Ελλάδα, δεν αναφέρεται στην έκθεση, αλλά το αναφέρω σαν παράδειγμα, όπου έχει από το 2007 υπογράψει ε, ε, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την Ανάπτυξη των Πρωτοβουλειών και μόλις πρόσφατα ενεργοποιήθηκαν αυτές οι διαδικασίες. λοιπόν εγρήγορση προσαρμοστικότητα και συντονισμός των απαραίτητων μέσων για την καλή αξιοποίηση της περιφερειακής πολιτικής. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό υποστηρίζω τις προτάσεις της ηγητρίας και από τη δική μου εμπειρία στη δική μου χώρα είδα τα πλεονεκτήματα όπως τα είδα και στο Μανχάιν πριν από δύο εβδομάδες τα θετικά στοιχεία προκύπτουν από αυτή τη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούν να βοηθηθούν ιδιαίτερα αυτέ οι περιοχέ. Η δική μου περιοχή πήρε μια χορήγηση για το επιχειρήν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να τονίσω ιδίω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η χρηματοδότηση και είχε σημαντικό αντίκτυπο εν γέννη στον κόσμο το να έχουμε καινοτόμους και αυτούς οι οποίοι μπορούν να προχωρήσουν σε επιχειρηματικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί μπορούν, λίγοι μπορούν να κάνουν καινοτομίε και πολλοί μπορούν να μιμηθούν μονάχα. Έχω δει λοιπόν αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι αυτά έχουν ευνοήσει όλες τις περιοχές μας, αλλά και με τη μιμητική μπορούν να ευνοηθούν και άλλες περιοχές δεν πρέπει λοιπόν το ΑΕΠ να είναι το μόνο στοιχείο με το οποίο καθορίζεται η αγοραστική δύναμη των περιοχών. Ευχαριστώ την κυρία εισηγήτρια και την συγχαίρω. Τη συγχαίρω για την εξαιρετική της εργασία. Όλοι γνωρίζουμε ότι η καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι κάτι το τελείως απαραίτητο και ότι η περιφερειακή διάσταση των αγών αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική όπως και στη στρατηγική για το 2020. Μέσα στα πλαίσια της τωρινής κρίσης είναι απαραίτητο να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για την χρήση των ταμείων συνοχής και για τα κριτήρια επιλογής των προγραμμάτων. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, δηλαδή ως προς την επίτευξη των στόχων μας. Νομίζω ότι στους βασικούς τομείς της οικονομίας πρέπει να υπάρξει μια εγγύηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής είναι απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μόνο έτσι θα καταλήξουμε σε βιώσιμη ανάπτυξη για το σύνολο της Ένωσης. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, θέλω να ευχαριστήσω την δυνατότητα να λάβω το λόγο παρά το γεγονό ότι είναι αργά πια το βράδυ. Η πολιτική συνοχή πολύ λίγε φορέ είχε τόσο μεγάλη σημασία όσο τώρα μέσα στα πλαίσια τη οικονομική κρίση. Είναι σαφέ ότι η κρίση οδηγεί σε απώλεια θέσεων απασχόληση που απαιτούνται Σημαντικέ επενδύσει από τα κράτη-μέλη για να ανακτήσουμε τι θέσει εργασία. Γι' αυτό πιστεύω πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στην πολιτική συνοχή να λειτουργήσει και στι περιφέρειε με επενδύσει. Χρειαζόμαστε όλα τα ευρώ τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει ιδιαίτερα στις περιοχές του στόχου 2 να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ποσά. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν σωστέ διαδικασίε για όλα αυτά, να υπάρχει μια αξιοπιστία και μια δυνατότητα σωστού σχεδιασμού, αλλά υπάρχουν και περιπτώσει όπω αυτή στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, όπου θα πρέπει να έχουμε και μια πραγματική ευελιξία. Διότι αυτή η ευελιξία θα μα βοηθήσει για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερε δυνατότητε στι περιφερειέ μα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σικέρσκι για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μπορέσει να ξεπεράσει την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Πρέπει πλέον να ξεπεράσουμε και τα διαφορετικά προβλήματα τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια μέσα από την κρίση αυτή. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει μια σειρά πρωτοβουλειών που θα μπορέσουν να οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη εκ νέου και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Θέλουμε να προωθήσουμε την καινοτομία, να δημιουργήσουμε νέες έξυπνες θέσεις απασχόλησης και να προχωρήσουμε και στον τομέα της πολιτική συνοχής θα πρέπει φυσικά όλα αυτά να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παρουσία των μέσων που έχουμε. Πρέπει να επενδύουμε τις ε, πιστώσεις που έχουμε στη διάθεσή μας με έξυπνο τρόπο για να οδηγήσουμε στη μεγαλύτερη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σεβόμενη την αρχή της αλληλεγγύης και σεβόμενη και την σωστή λειτουργία και εύρεθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε αποσπασματικά, δεν μπορούμε να ασχολείται ο καθένας μόνο με το δικό του περιβολάκι, αλλά θα πρέπει όλοι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δουλέψουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση των κρατών μελών βρίσκονται σε μια διαδικασία εφαρμογής σκληρών μέτρων για να μπορέσει να υπάρχει ανάκαμψη των οικονομιών των κρατών μέρων. Πέραν των μέτρων λιτότητας που έχουν εγκριθεί, πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε να κάνουμε και επενδύσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δεύτερος στόχος της πολιτικής συνοχής είναι να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και να απασχολήσουμε και περισσότερους ανθρώπους. Η πολιτική λοιπόν αυτή θα πρέπει να εξυπηρετήσει και την καλύτερη σύγκληση των χωρών μέρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για τη χώρα μου ένας τρόπος εξόδου από την κρίση είναι να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενθαρρυνθούν οι τοπικές αρχές να προχωρήσουν σε σχέδια με υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Κύριε Σεσκοβίτς, από... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια και αντιπρόεδρο για την έκθεσή της που αφορά το ρόλο της πολιτικής συνοχής στο σχέδιο και περαιτέρω. Η πολιτική συνοχής θεωρείται ως πολιτική στήριξης της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων και την επίτευξη πραγματικής σύγκλησης μέσω διαρθρωτικών αλλαγών. Με 347 δισεκατομμύρια για περίοδο από το 7 μέχρι το 13, 228 έχουν διατεθεί ακριβώς για στόχους συνοχής και για δημόσιες επενδύσεις και για οικονομική πειθαρχία, δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν πρόκειται για πολιτική που αντιμετωπίζει τις κυκλικές κρίσεις, αντικυκλική πολιτική δηλαδή, αλλά για πραγματική επένδυση στην ανάπτυξη. Και τη θεωρούμε ως ένα σημείο κλειδί, ένα τμήμα κλειδί για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Αναθέρμανσης με κύριο στόχο την αντιμετώπιση των περισσότερων ή σημαντικότερων αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης. Γι' αυτό κάναμε συστάσεις και προτείναμε νομοσχέδια. Με δεύτερο στόχο την επιτάχυνση της χρηματοδότησης των ε, σχεδίων που έχουν ήδη εγκριθεί για αυτές τις δημοσιονομικές προοπτικές μέσω αυξημένης προχρηματοδότησης και μέτρων απλοποίησης. Οι νομοθετικές αυτές αλλαγές άρχισαν από τον Απρίλιο του 9 και οι ανακοινώσεις της Επιτροπής ενεκρίθησαν προηγουμένως από το Δεκέμβριο του 8. Η νομοθετική αυτή δέσμη λοιπόν έχει εγκριθεί συνολικά μέσα σε πέντε μήνες, πράγμα το οποίο συμβαδίζει απόλυτα με την αναγκαιότητα ταχείας αντιμετώπισης. Θα ήθελα να τονίσω κύριε Πρόεδρε ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται και στην ποιότητα της διαθεσμικής συνεργασίας, ιδιαίτερα δε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί συμφωνούσατε και εσείς να υπάρξει μία σύντομη αντιμετώπιση. Γενικά τα μέτρα αυτά θεωρήθηκαν θετικά αντιμετώπιση του προβλήματος της επιτάχυνσης των επενδύσεων και ήταν ταυτόχρονα επαρκώς ευέλικτα ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τους στόχους που τα βόλευαν καλύτερα ανάλογα με τις περιφερειακές τους ανάγκες, δεν ήταν μονολυθικά. Επίσης συνέβαλαν στη βελτίωση των, της εφαρμογής των νομοσχεδίων και των προγραμμάτων που αφορούν την πολιτική συνοχής μέσω καλύτερης διαχείρισης. Και δεν στόχευαν μόνο στην καταπολέμηση της κρίσης, αλλά και στην αναθέρμανση μετά την κρίση. Τέλος, η Κομισιόν θα παρουσιάσει έκθεση ως προς την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της επιπτώσεις των μέτρων εφόσον έχει υποσχεθεί κάτι τέτοιο ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμως. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Αγαπητοί συνάδελφοι, η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθεί αύριο, 3η 6 Ιουλίου 2010, από τις 9 ως τις 13, από τις 15 ως τις 20 και 30 και από τις 21 μέχρι τις 24. Η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνεδρίαση έληξε. Καληνύχτα σε όλους.